Παρακαλώ κύριε Κοφεράτη. Και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί ούτε η δική μου συσκευή. Παρακαλώ να καταγράψετε και τη δική μου τη ψήφο. Ε, θα ληφθεί αυτό υπόψη από τι αρμόδιε υπηρεσίε. Τώρα λοιπόν η Μέση Διάταξη προβλέπει την ψηφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση του κυρίου Τικάου σχετικά με τι κυρίε Τικάου, με συγχωρείτε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα και τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Βραζιλία σχετικά με τι ορισμένε πτυχέ των αεροπορικών μεταφορών. Ε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται έκθεση Βαντεκάμπ με βάση τη μερίσια διάταξη η ίδια ε, διαδικασία για την ε, ψηφοφορία ε, αφορά στην συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Ισλανδίας του Βασιλείου της Νορβηγίας Ελβετικής Ομοσπονδίας και του Πληκάτου του Λίχτενστάιν υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται έκθεση Κοέλιο ίδια διαδικασία για την προσχώρηση του Λίχτενστάιν στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές η έκθεση εγκρίνεται. Η Μέση Διάταξη προβλέπει την ψηφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση του Σαντέλφ κ. Χούλμαια για την ε, προσχώρηση του Λίχτενστάιν στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία ε, ε, σχετικά με τον προσδιορισμό που είναι υπέρ, του κράτου που είναι υπεύθυνο για την του ασύλου υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση του κυρίου Μακοβέη για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Βραζιλία σχετικά με την εξαίρεση από την υποχρέωση τη βραχία διαμονή για του κατόχου κοινών διαβατηρίων. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, παρακαλώ, εγκρίνεται. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση του κυρίου Έντσου σχετικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση βραχία διαμόνηση για του πραγματικών υπηρεσιακών ή επίσημων διαβατηρίων. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία με την ίδια διαδικασία για την έκθεση της ε, κυρίας Γκέιπχατ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία για την έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και Πούλμαν. Ε, εισηγητή ο κύριος Καμτσάν. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, και το δικό μου μηχάνημα α, ε, δεν λειτουργεί. E Εντάξει λοιπόν, θα ληφθεί υπόψη τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία για την έκθεση. Παρακαλώ, κύριο Αλφάνο. Η κυρία Αλφάνο, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Χτε έχασα την κάρτα μου κάπου εκεί στην Επιτροπή και την ψάχνω, την βρω. Παρακαλώ να δηλώσετε ότι, να καταγράψετε ότι ψήφισα αποχή για την έκθεση Καντσάμ. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ε, θα καταγραφεί τώρα, προβλέπεται η ε, ψηφορία της έκθεσης Κάλαναν ε, σχετικά με τις εκπομπές καυσερίων από καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν το υπαριθμόν 1 σε ξεχωριστές ψηφορίες. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφορία για το πρώτο, πρίμα, πρώτο τμήμα. Με ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση της Επιτροπής ως τροποποιήθηκε ε, με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ε, για την πρόταση ψηφίσματος, σχέδιο ψηφίσματος, με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε η έκθεση συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Λένε σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ψηφίζουμε παρακαλώ με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίθηκε η έκθεση. Η σε διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία για την έκθεση ε, του κυρίου Μπελέ ε, σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Κύριε Σιλβέστρη, Πρόεδρε, εγώ κατά λάθο ε, υπερψήφισα, αλλά η δική μου η για την προηγούμενη ε, ψηφορία ήταν κατά, παρακαλώ να το καταγράψετε. Εντάξει, λαμβάνετε υπόψη. Καταγράφηκε, λέει η Πρόεδρος. Τώρα λοιπόν προχωράμε. Μισό λεπτό. Ο κύριος Πιτέλα. Θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ κατά λάθο υπερψήφισα, αλλά ήθελα να δηλώσω αποχή παρακαλώ. Eh, Prego, Presidente. Prego. Presidente. Basta. Sí. Errore en la votación, mi voto. Εγώ έκανα λάθος στην ψηφοφορία, είμαι κατά. Prego, Presidente Aguiar. Sí, señora. Ο κύριος η ψηφοφορία έγινε πολύ κοντά στην προηγούμενη και εγώ είμαι κατά. Δεν πρόλαβα να ψηφίσω καν, αλλά είμαι κατά. Έγιναν ε, πολύ απανοτά οι δύο ψηφοφορίες και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα τεχνίας περιμένει, περιμένει την ε, επίλυση κρεμοδικίας ε, στο δικαστήριο για μια απόφαση που αναμένουμε στις 8 Μαρτίου. Γι' αυτό προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία μέχρι ότου αποφαθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα δικαιοδοσία ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώ. Κύριε Σιλβέστρη, ε, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση της έκθεσης Μπελέτ. Ψηφίζουμε λοιπόν για την τροπολογία υπερθυμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Παρακαλώ να σηκώστε το χέρι. Κατά αποχές ε, πρέπει να επαληθεύσουμε γιατί δεν σηκώσετε καλά τα χέρια σας. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Προφανώς, ε, σαφέστατα, απορρίπτεται η τροπολογία. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία υπερθυμών 32. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 τροπολογίες ε, της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας. Ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Μπελέτ ε, προτείνει μια προφορική τροπολογία. Όχι, κατέπεσε. Όχι, όχι, δεν κατέπεσε. Την ε, καταθέτει την προφορική τροπολογία ε, στην υπαριθμόν 33, ως εκ τούτου του δίνω το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφορική τροπολογία για την αποζημίωση αγροτών και ευχαριστώ την κυρία Ριβαζή για την πρωτοβουλία της και έχει ως εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μέχρι το Μάρτιο του 2012 μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη σκοπιμότητα μηχανισμού αποζημίωσης αγροτών των οποίων οι ζωοτροφές ε, μολύνθηκαν πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα και δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά. Και ο μηχανισμός να βασίζεται στην αρχή ενών πληρώνει και αν χρειαστεί να συνοδευτεί και από νομοθετική πρόταση έκθεση που να ιδρύει αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κοινή πρόταση πέντε πολιτικών ομάδων. Δε. Πολύ ωραία. Αντιρρήσει, παρακαλώ. Ε, υπάρχουν, υπάρχει κανεί που να διαφωνεί σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 33. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση της Επιτροπής ως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση. Ψηφίζουμε για το σχέδιο ψηφίσματος, νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα λοιπόν ξεκινάμε με τις επεξηγήσεις ψήφου.